του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε σχέση με, το, με την ασυλία του κυρίου Λουίτζι Μπέρλιγκουερ ζήτησαν να επιβεβαιωθούν τα προνόμια και η ασυλία.